Πολλοί από εσά θα πρέπει να φροντίσουμε να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους στο γεωργικό τομέα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνει η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Η επόμενη Ολομέλεια, Τρίτη, 18 Ιανουαρίου, από τις 9 στη 1, από τις 3 στις 8 και από τις 9 στις 12 τα μεσάνυχτα. Η ημερήσια διάταξη την έχετε και στην ιστοσελίδα. Πέρα στις σας.